Αν επιτρέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Παρακαλώ. Οι συνάδελφοι από τα Εθνικά αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθίστε, θέλουμε να ξεκινήσουμε. Είναι πολύ δύσκολο να αρχίσει η συζήτηση όσο εσείς κυκλοφορείτε στο ημικύκλιο. Καθίστε παρακαλώ. Θα ήθελα από την αρχή να επισημάνω πριν ξεκινήσουμε ότι προβλέπεται η διερμηνία σε πολλές γλώσσες. Πλην μία σε ξεσονορίζω. Όλες οι γλώσσες λοιπόν είναι διαθέσιμες αρκεί να επιλέξετε το κατάλληλο κανάλι που προβλέπετε για την επιλογή της γλώσσας. Έχετε επίσης και πλήρη τεκμηρίωση για την διαδικασία της Στοκχόλμης και τα έγγραφα που βρίσκονται έξω από το ημικύκλιο. Πρόκειται για τεκμηρίωση την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον στον τομέα αυτών. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάτε να πάρετε τα έγγραφα αν όχι τώρα, πάντως αργότερα. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, αγαπητή συνεδρίαση, αγαπητή συνεδρία, ε, αγαπητή συνάδελφη, ξεκινώ καλωσορίζοντά σα όλους, αλλά κυρίω τον κύριο Πέρλ Βέστερμπεργκ που βρίσκεται στα αριστερά μου. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ρίξτακ, του Σουηδικού Κοινοβουλίου, ο οποίος θα συμπροεδρεύσει μαζί μου και στις δύο ημέρες αυτές τον τη συνεδρίασή μα με το Εθνικό Κοινοβούλια, των οποίων και ευχαριστώ και για τι προσπαθίε του στην προετοιμασία τη ε, συνεδρίαση. Το προσωπικό του, όπως και το δικό μας προσωπικό, συνεργάστηκαν στενά στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ όλους όσοι μόχθησαν για την προετοιμασία αυτής της ε, συνεδρίασης και επίσης θα ήθελα πολύ θερμά να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών, αλλά και από τα Κοινοβούλια των Υποψηφίων Κρατών. Τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε. Και εσείς είστε οικοδεσπότες αυτής εδώ της συνεδρίασης. Ιδιαιτέρως δε θα αναφερθώ στον κύριο Χουάν Φερνάντο Λόμπες Ακριλιάς, πρόεδρο της ε, Επιτροπής των Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ε, και Ευρωβουλευτή φυσικά, ο οποίος θα αναλάβει να κάνει την αρχική εισήγηση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκ μέρους δε του Σουηδικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Τόμας Μπόκστρουμ, μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, θεμάτων δικαιοσύνης, νομικών θυμάτων της Ρίξτακ, θα κάνει και αυτός με την πλευρά του κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Επίσης, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να καλωσορίσω εδώ εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Λουκ Φαντερβάντεν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, από, και εκπρόσωπο της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλους, όλοι δε οι λοιποί προσκεκλημένοι επίσης, καλώς ήρθατε. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι έχετε φορέσει τα ακουστικά σας και έτσι μπορώ να ε, αλλάξω γλώσσα και να μιλήσω πολωνικά. Πρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε σε αυτήν την πρώτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Ήταν πάντα σημαντική η συνεργασία μας η συνεργασία μεταξύ Εθνικού και Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε συνεργασία μέσω της ΚΟΖΑΚ ε, που ήδη αριθμεί 20 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, Έξι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζουν σε μια κοινή συνεδρία στην οποία συμμετέχουν από κάθε κράτος μέλη έξι εθνικοί βουλευτές μέσα στην ΚΟΖΑΚ. Έχουμε επίσης τη διάσκεψη των Προέδρων των Εθνικών Κοινοβουλίων και πιο πρόσφατα έχουμε εισαγάγει νέα μέσα και όργανα για να διευκολύνουμε την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια στιγμή πολύ ουσιαστική τη συνεδρίασή μας, μια κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια. Η συνθήκη της Λισαβόνας από Δίδη προβλέπει δραστήριο ρόλο για τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τη θέση της ισχύ σε δύο-τρεις εβδομάδες ακόμη, δηλαδή από 1η ε, Δεκεμβρίου, μπορούμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικά την συνεργασία. Με την διακοινοβουλευτική αυτή συνεδρίαση νομίζω ότι μπορούμε ήδη να συστήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Η Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Συνόδου για δε τους συμπολίτε μας τα ζητήματα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας ε, που είναι πολύ σημαντικά πρέπει να συζητηθούν και όταν τεθεί σε ισχύ η νέα συνθήκη θα έχουμε και νέους τομείς συνεργασίας όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς από πλευρά σας, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα είστε σε θέση να επαληθεύετε κάθε νομοθετικό κείμενο που προτείνεται υπό το πρίσμα της επικουρικότητας, υπό τον όρο της επικουρικότητας και θα διατυπώνει τις γνωμοδοτήσεις σας. Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα ακόμη σκοπεύει να εισαγάγει τη σχετική τροποποίηση στον κανονισμό του για να προχωρήσει το χέτερο δυνατό στη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Παρακαλώ λοιπόν έχετε υπόψη ότι κάθε νομοθέτημα που πρόκειται να ε, εξεταστεί υπό αυτό το πρίσμα της ε, επικουρικότητας πρέπει να ε, πρέπει να περάσει από όλη τη δικασία αυτή του ελέγχου μέσα σε 8 εβδομάδες. Πρέπει επομένω να οργανώσουμε πολύ καλά και να συγχρονίσουμε πολύ καλά τι εργασίε μα για να είμαστε αποτελεσματικοί και ταχύρυθμοι. Το Κοινοβούλιο με, τη, με το Προεδρείο του και τη, τη Γενική του Γραμματεία ήδη ξεκινά κάποιε προσπάθειε πρακτικέ έτσι ώστε στο νέο αυτό τομέα συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δηλαδή να έχουμε άμεση συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλευτικών μα επιτροπών ένα τομέα από τον ε, στον οποίο έχουμε στρίξει πολλές ελπίδες. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ξεκινούμε με τα θέματα της Europol και της Eurojust. Αυτά θα είναι, νομίζουμε, και το δοκιμαστήριο ηλδία λίθος της συνεργασίας μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε την ΚΟΖΑΚ ως ε, χώρο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Έχουμε κοινέ διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις όπως η σημερινή μας και τώρα ξεκινάμε με μια τρίτη μορφή συνεργασίας στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και για να προχωρήσω τώρα στην σημερινή ημερήσια διάταξη, αυτά που έχουμε να συζητήσουμε μαζί με την ε, Σουηδική Προεδρία. Έχουμε ετοιμάσει τη θεματολογία μας για νέες κατευθυντήριες γραμμές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ε, τομέα της, του κοινοβουλευτικού ελέγχου, της κοινοβουλευτικής επαλήθευσης για την δικαιοσύνη και, την, ε, και τα εσωτερικά. Και με την συνεδρίαση του Φεβρουαρίου εφέτος στο Παρίσι υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή από το Συμβούλιο. Παραλαμβάνω ότι είμαστε ευγνώμονε προς τη Σουηδική Προεδρία η οποία ε, και, με την, και από την πλευρά τη υπεστήριξε την πρόταση αυτή και συνέχισε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό και περιμένουμε βεβαίω και τις προτάσεις των ε, εκπροσώπων και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για να κλείσω τις ε, παρατηρήσεις μου, πριν πάρει το λόγο ο κύριος και ο κύριο συμπρόεδρο. ε, ίσως θα έπρεπε να του δώσω πρώτα το λόγο για να μας δώσει και εκείνο τι δικέ του ιδέε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, ε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω από όλη την Ευρώπη σε αυτή την ε, κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση. Θα συζητήσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση της ε, ε, μελλοντικής πολιτικής ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το λεγόμενο πρόγραμμα Στοκχόλμης. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για την ασθενή και πολύ υποφελή συνεργασία εν ώψη της προετοιμασίας της κοινή αυτής κοινοβουλευτικής συνάντησης. Η διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και πιο σημαντική και λειτουργεί μέσα σε διάφορα πλαίσια, στα πλαίσια της ΚΟΖΑ και σε δια, πλαίσια διάφορων διασκέψεων. Πριν από 20 χρόνια, το 89, η ΚΟΖΑΚ συναντήθηκε για πρώτη φορά τα εθνικά κοινοβούλια συνεισφέρουν ενεργά στην καλή λειτουργία και στην αύξηση της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, εθνικά κοινοβούλια είμαστε ενεργοί εταίροι για να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα καλύτερα δυνατά. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά εισάγεται λοιπόν ε, στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ε, προβλέπονται έξι διάφοροι, διαφορετικοί τρόποι με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια ε, συνεισφέρουν ενεργά στην, σε μια εύρυθμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον τομέα της ελευθερίας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ούτω ώστε να συνεισφέρουν στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθώντας, ε, αξιολογώντας ε, τις ε, κοινοβουλευτικές πολιτικές και συμμετέχοντας στην αξιολόγηση της Eurojust καθώς και στην, στον πολιτικό έλεγχο και παρακολούθηση της Europol. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτό το τομέα θα καθοριστεί μέσα σε, κάποια, σε κάποιους κανονισμούς που θα υιοθετηθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ο βασικός σκοπός αυτός, αυτών των κανονισμών είναι να καθοριστεί ο, ο τρόπος εργασίας και οι δομές, το πεδίο εργασιών και οι εργασίες της Eurojust και Europol. Τα συμπεράσματα της διάσκεψης των Προέδρων του Κοινοβουλίου στο Παρίσι πριν από λίγο καιρό τόνισαν το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων για να δημιουργηθούν νέες προτεραιότητες για μια ευρωπαϊκή δράση για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικοδόμησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η συνέχιση των ε, συμπερασμάτων ε, της διάσκεψης ε, των Προέδρων επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε σε καθημερινή βάση με τους βουλευτές, οδήγησαν σε αυτή την κοινή κοινοβουλευτική συνάντηση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, κάποιοι τομείς ήδη έχουν υπογραμμιστεί σε δύο από τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν. Την συνάντηση της ΚΟΖΑΚ 4 με 6 Οκτωβρίου που ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Η διακοινοβουλευτική συνάντηση 11 και 12 Οκτωβρίου εξέτασε το θέμα της ισορροπημένης προσέγγισης στη νομική ασφάλεια και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορία των ανθρώπων. Το να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των πολιτών ήταν ο τίτλος αυτής της συνάντησης. Και τα θέματα στην περίσσια διάταξη τονίζουν κάποια από τα ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε τα επόμενα χρόνια, 2010 ε, με 2014. Επίσης θα πρέπει να εισαχθούν και νέες μέθοδοι εργασίας. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη ε, της Ισουηδίας θα σας εξηγήσει πώς ε, θα αντιμετωπίσει το νέο πολιτέ πρόγραμμα της Νέα Προκλήση. Ακόμα μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους σας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. κύριε Βέστερμπεργκε, πρόεδρε του Σουηδικού Κοινοβουλίου, για τα εισαγωγικά σας λόγια. Όπως είπαμε, συμπροεδρεύουμε σε αυτή την συνάντηση μαζί με τον κύριο Βέστερμπεργκ. Θα του δώσω τώρα το λόγο για να προεδρεύσει αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λόπες Αγουιλάρ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο κύριε Λόπες Αγουιλάρ για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Bonjour à tous. Good afternoon. Είναι μεγάλη χαρά που έχω τη δυνατότητα να πάρω το λόγο σε αυτήν την κοινή συνάντηση των μελών των κοινοβουλίων των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι τιμή μου που παίρνω το λόγο σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών υπεύθυνη επίσης και για τα θέματα δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. Και θα σας μιλήσω, θα σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία από τη δουλειά την οποία έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών τις τελευταίες εβδομάδες. γύρω από την προσπάθεια προσαρμογής του προγράμματος της Στοκόλμης είναι θα έλεγα τα μέτρα που τίνουν στην ανάπτυξη ενός κοινού χώρου ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα μου επιτρέψετε τώρα να χρησιμοποιήσω την ισπανική μητρική μου γλώσσα για να μοιραστώ καλύτερα αυτό το προσχέδιο θα έλεγα περιγραφής του τι έχει γίνει μέχρι τώρα, κυρίως όμως της προσπάθειας η οποία μένει ακόμα να αναλυφθεί στις επόμενες εβδομάδες και που έχει σαν στόχο να προχωρήσουμε στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης και να προχωρήσουμε στην τελική αποδοχή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10 η Δεκεμβρίου, όπως επίσης και της υιοθέτηση του προγράμματος δράσης από την επόμενη, ε, επερχόμενη θα έλεγα, Ισπανική Προεδρία μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το πόσο είναι σημαντική για μένα αυτή η τόσο συμβολική στιγμή όπου παίρνει περιεχόμενο η πολιτική της και η συνταγματική της Πρόκειται λοιπόν για ένα δείγμα πολιτισμού που καθιστά ξεχωριστή την Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Μιλάμε για υπηκότητα, μιλάμε για κοινέ συνταγματικέ παραδόσεις, για σύγκληση ελευθερίας και ασφάλειας που αποτελούν και την σπονδυλική στήλη αυτής της ε, εκπολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή της σύλληψής της ως ιδέα. Σε δύο εβδομάδες, δηλαδή αρκετά σύντομα, θα αρχίσει τελικά να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας που θα αποτελέσει μια ιστορική ευκαιρία να ξεπεράσουμε τη συνταγματική συζήτηση αυτή που κράτησε τουλάχιστον 10 χρόνια η οποία έφαγε πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ δουλειά, ουσιαστικό χρόνο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση αλλά πρόκειται για χρόνο ο οποίος επενδύθηκε σωστά αν δηλαδή εμείς μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτό το όραμα για την υπηκότητα, για το ευρωπαϊκό ανήκειν. Εμείς είμαστε βουλευτές, είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να εκπροσωπούμε τους πολίτες και απέναντι στους πολίτες εμείς ε, είμαστε υπόχρεοι και με τη δουλειά μας και με αυτά που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάστηκαν οι Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών Συνταγματικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης με τις ομόλογες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων για να μπορέσουν ακριβώς να υπογραμμίσουν το πόσο θα πρέπει εμείς να τονίσουμε την όλη διεργασία της Στοκχόλμης. Αυτό έγινε τότε και με το πρόγραμμα του Τάμπερε υπό Φιλανδική Προεδρία. Είχαμε δηλαδή μία πολυετή ατζέντα που μπόρεσε να δώσει περιεχόμενο στην συνθήκη του Άμστερνταμ στην έννοια της ελευθερίας και της ασφάλειας. Μετά είχαμε την ατζέντα της Χάγης το 2004 και η Σουηδική Προεδρία κατέβαλε την προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει μια νέα προπτική στο χώρο δικαιοσύνης και ελευθερίας με την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που αποτελεί ένα άλμα προς τα διότι ακριβώς κλείνει αυτή τη δεκαετή συνταγματική συζήτηση διότι ιδρύεται αυτή η αρχή του πολίτη της υπηκότητας της Ευρώπης και δίνεται και η νομοθετική διάσταση, το νομικό πλαίσιο αυτού του καθεστώτος και μειώνεται η απόσταση μεταξύ του πρώτου πυλώνα και του τρίτου πυλώνα μεταξύ των οποίων εμείς κινηθήκαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα είναι λοιπόν συναποφασιστής ε, το Κοινοβούλιο μαζί με το εκτελεστικό όργανο και θα εμπλέκει και τα εθνικά κοινοβούλια για να ενισχυθεί αυτή η συμμερισμένη ιδιότητα του πολίτη. Έτσι τονίζεται και το δεύτερο άρθρο της Λισαβόνας που μιλάει για τον πλουραλισμό, ανεκτικότητα, δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων, ισονομία, ε, χωρίς καμία διάκριση σε καμία από αυτές τις θεωρήσεις. Οι Ευρωπαίοι πολίτες λοιπόν θα είναι και πρωταγωνιστές της νομιμοποίησης αυτών των δικαιωμάτων αλλά και δικαιούχοι ταυτόχρονα. Χρειάζεται λοιπόν συνεχής και καρποφόρος διάλογος μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναλογικότητα και την επικουρικότητα μέσα από το τις οποίες θα πρέπει να διέπεται αυτός ο νομοθετικός διάλογος μεταξύ των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο χώρο της ελευθερίας ασφάλειας δικαιοσύνης. Η δημοκρατική ασφάλεια θα πρέπει να διέπει την όλη νομοθετική διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε ασάφεια ή αμφισημία οποιαδήποτε αντίφαση ή επικάλυψη ως προς την νομοθετική προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτό βγήκε από τις κοινέ συνεδριάσεις των επιτροπών μας, δικαιοσύνη συνταγματικών υποθέσεων, και δημοσίων ελευθεριών για να συζητηθεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Συμπορευθήκαμε λοιπόν τρεις συζητητές για την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων ο κύριος Κάρλο Κασίνη για τις νομικές υποθέσεις ο Λουίτζι Μπερλιγκουέρ και για ο υποφαινόμενος ως πρόεδρος της Επιτροπής Λίμπε. Εργαστήκαμε και συντάξαμε ένα κοινό ψήφισμα που καλεί σε μία προσπάθεια για την ομοθετική ποιότητα, αποτελεσματικότητα, ισότητα και δικαιοσύνη που είναι και πρωταρχικός στόχος αυτού του που λιετούς προγράμματος, πέντα ε, πενταετούς, γιατί είναι τα πέντε επόμενα χρόνια που θα εγκριθούν το Δεκέμβριο στην Στοκχόλμη από τη Σουηδική Προεδρία. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει προωθήσει η Σουηδική Προεδρία είναι πολύ φιλόδοξο και θα αποτελέσει τον κορμό της αρχής του πολίτη, της υπηκότητας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Η ε, εξωτερικά σύνορα. Ε, συνεργασία δικαιοσύνη και αστική συνεργασία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας, την ασφάλεια στην διακίνηση, συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για να καταπολεμήσουμε και το οργανωμένο έγκλημα και την, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και της τρομοκρατίας. Όλες αυτές οι απειλές είναι πραγματικές και απαιτούν προσπάθεια χρονοβόρα και που ξεφεύγει από τις ατομικές προσπάθειες του καθένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν δίνουν απαλλαγή στα κράτη-μέλη και στο ρόλο που πρέπει αυτά να παίξουν. Χρειάζεται λοιπόν ευφύς διάλογος, συνεργασία, ποιότητα μεταξύ των νομοθετικών μας οργάνων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι λοιπόν αυτό αφορά την δική μας κοινωνία των πολιτών στο να αναλαμβάνει πρωτοβουλία διότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει το χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου έχουμε νομική προστασία κατά των καταχρήσεων και των αδικιών όπως ποτέ δεν συνέβη στην ιστορία της Ένωσης. Έχουμε λοιπόν μία πορεία που σίγουρα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στη φάση της προσαρμογής διότι όλο το κοινοτικό και εκτιμένο των τελευταίων δέκα ετών από το Τάμπερε και μετά θα πρέπει να μεταφερθεί μετά από μια μεταβατική περίοδο να εφαρμοστεί η, η προσαρμογή όλων των νομοθετικών προϊόντων, νομοθετικών παραγόγων του τρίτου πυλώνα στη νέα κατάσταση πρέπει να αλλάξει, χρειάζεται συμπλήρωμα. Χρειάζεται μια λισαβονοποίηση και αυτό θα απαιτήσει σκληρή εργασία από όλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται αιμονή, προσοχή, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν έγκαιρα. τον Ιούνιο του 2010 υπό Ισπανική Προεδρία θα έχουμε μια νέα ουσιαστική στιγμή ολοκλήρωσης των αρχών της Στοκχόλμης διότι οι πολίτες ατενίζουν προς εμάς, έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτήν την προσπάθεια που θα μοιραστούμε. Θα υποβληθεί στην Ολομέλεια αυτό το κοινό ψήφισμα και σας το λέω προκαταβολικά ότι έχουμε την καλύτερη διάθεση ούτως ώστε να δεχθούμε ό,τι τροποποίησεις θελήσετε και συνεισφέρετε κατά τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που μπόρεσα να έρθω σήμερα στις Βρυξέλλες εδώ για να σας μιλήσω για τα θέματα αυτά. Το θέμα μας είναι Ευρώπη για τους πολίτες. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα επαρκώς σοβαρό για να μαζευόμαστε εδώ όλοι οι βουλευτές να συζητήσουμε τέτοια μεγαλόπνοα θέματα ελπίζοντας ότι αυτή η συνεδρίαση θα μας οδηγήσει σε αποτελέσματα. Οι βουλευτές, άνδρες και γυναίκες, έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να παίξουμε όταν πρέπει να επηρεάσουμε τις κυβερνήσεις μας. σε θέματα εσωτερικών υποθέσεων τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, θα αρχίσει σύντομα να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και θα αρχίσει να αλλάζει και ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων. Διότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στην καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών πολλά πράγματα θα αλλάξουν και στα εθνικά κοινοβούλια θα αλλάξουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι στο παρελθόν στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ομιμότητά μας στα μάτια των πολιτών. Η ευρωπαϊκή συνεργασία τα τελευταία χρόνια αύξησε τη σημασία της. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Υπάρχει μια μεγάλη συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για την συνεργασία ώστε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Στον ποινικό τομέα ενισχύθηκε η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή οι αστυνομίες ενός κράτους μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από άλλες αστυνομίες χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια. Όλα αυτά λοιπόν διευκόλυναν τις διαδικασίες ούτως ώστε να έχουμε τη μια σχετικά εύκολη διαδικασία έκδοσης των διαφόρων εγκληματιών από τη μια χώρα στην, από μια χώρα άλλη. Θα εγκριθεί λοιπόν το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η καταπολέμηση του εγκλήματος είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί όμως κάτι τέτοιο να μη συμπορεύεται και με την εγγύηση των ατομικών δικαιωμάτων. Εμείς οι βουλευτές θα έχουμε την εντολή να συμμετέχουμε σε αυτές τις εργασίες και να ενημερώνουμε τους πολίτες μας σχετικά. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα εγκριθεί τον Δεκέμβριο και αυτή τη στιγμή εγκριθεί το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα πρέπει να ξεκινήσουμε την επεξεργασία του, τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα πρέπει να αναλάβουμε ούτως ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Όπως επίσης να δούμε και με το τι τρόπο θα προσεγγίσουμε αυτούς τους στόχους για να βελτιώσουμε και την νομική ασφάλεια των πολιτών αλλά και για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Χρειάζονται λοιπόν αηφόρες λύσεις. Εγώ προσδοκώ ιδιαίτερα στις συζητήσεις που θα γίνουν εδώ και ελπίζω ότι θα έχουμε μία συζήτηση ανοιχτή και διαφανή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα θα ήθελα να πούμε ότι αρχίζουμε τη συζήτηση, το διάλογο. Θα το επαναλάβω, ασφαλώς θα γνωρίζετε πώς ε, ε, λειτουργεί αυτός ο διάλογος, αλλά θα επαναλάβω τους κανόνες. Έχουμε καταρχάς τους ε, βουλευτές που θέλουν να παρεύουν στην συζήτηση, τους οποίους παρακαλούμε να συμπληρώσουν το φυλάδιο, το κίτρινο φυλάδιο που ε, συνεπάγεται έτοιμα η χρόνου ομιλίας για τη Δευτέρα. Το έχουν λάβει ήδη οι αντιπροσωπείες. Το κίτρινο φυλάδιο μέσα στους φακέλους σας. Είναι μια σελίδα χαρτί κίτρινη. Και θα συμπληρώσουμε ανάλογα τον κατάλογο των αγορητών με την συνεργασία της γραμματείας. Οι κανόνες. Τέσσερα μία Πρώτον, ε, έχουμε την ακολουθία. Δύο από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν επιστρέψει δηλαδή ευκαιρίε να λάβουν τον λόγο οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Χρόνο ομιλία τρία λεπτά για κάθε παρέμβαση. Θα τον βλέπετε άλλωστε στην οθόνη. Ε, δυνατότητα χρήση ε, του λεγόμενου γαλάζιου δελτίου καινούρια διαδικασία στο κοινοβούλιο μας με μέγιστο 30 δευτερόλεπτα για κάθε ερώτηση που ενδεχομένως, τέταρτο σημείο, θέλετε να διατυπώσετε προς οποιονδήποτε ομιλητή. Η ερώτηση προς οποιοδήποτε ομιλητή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κάνετε σήμα με το γαλάζιο αυτό δελτίο και σας δίνεται η ευκαιρία για 30 δευτερόλεπτα να διατυπώσετε την ερώτησή σας. Και επίσης για την απάντησή σε αυτήν θα έχετε 30 δευτερόλεπτα. Θα έχει 30 δευτερόλεπτα ο εν λόγω ομιλητής να απαντήσει. Οι δύο δε συμπρόεδροι αποφασίζουμε εάν υπάρξει αν ε, ε, όντω είναι δυνατή η χρήση αυτή τη διαδικασία του γαλάζιου δηλητηρίου. Γιατί αν δούμε ότι γίνονται συνεχεί διακοπέ με πολλέ ερωτήσει, προφανώ δεν θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διαδικασία. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε και όλους, θα έχουν, όλους όσοι θα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των αγορητών. Αναλόγω λοιπόν, εάν είναι πολλέ, υπερβολικά πολλέ ερωτήσει, γιατί όπω είπα, ο καθένα μπορεί να διακόπτει ε, για κάθε θέμα. Έχω λοιπόν δύο γαλάζια δελτία. Η κυρία Κόριαν Γιόνκερ από την κοινοβουλευτική συνέρευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια βουλευτής από τις κάτω χώρες, η οποία θα λάβει το χώρο. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται να έρθετε εδώ. Από, την παρέ... από το κάθισμά σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Εκεί είστε μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Σουηδικό Ρίξτακ ε, που προσκάλεσαν την ε, αντιπροσωπεία τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, Να ε, χαιρετήσω και τον κύριο Αγγιλάρ, πρώην συνάδελφο, γιατί ήταν στο Συμβούλιο τη Ευρώπη πριν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σα ευχαριστούμε που μα δίνετε την ευκαιρία συμμετάσχοντα σε αυτή τη συνεδρία τη 20 του να συμβάλλουμε και εμεί στην ολοκλήρωση τη διαδικασία, του εγγράφου τη της τη τη οποία αντίκτυπο θα δουν όχι μόνο το κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα θα έχει ένα φαινόμενο ομόκεντρων κύκλων σε μια πέτρα που πέφτει σε βαλτόδι νερά και θα επηρεάσει όλα τα κράτη και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι φιλόδοξη αυτή η διαδικασία και προβάλλει πολλά από τα θέματα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο τη θέλουμε πολύ σημαντική και θέλουμε να καταγραφεί απολύτω και διεξοδικά το έργο της έτσι ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια δουλειά αργότερα. Επίσης με χαρά σημειώνω το σχέδιο προγράμματος ε, καταγράφει κάποιες από τις προσπάθειες που έχει ήδη ολοκληρώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη δυνατότητα να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης περαιτέρω εξελίξεις. Πλην όμως περαιτέρω ε, ανάδειξη του ρόλου του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, την παρακολούθηση, την συνεργασία, την πολιτική σύμπραξη, νομίζω θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο να αναδείξουμε και επιπλέον να αναφερθούμε και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη οποία ε, το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αναδειχθεί στο πλαίσιο τη συνεργασία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, θα πρέπει να υποβάλω με χωριστό έγγραφο μια σειρά προτινόμενων τροπολογιών για το σχέδιο τη ε, Στοκχόλμη που προτείνουμε με βάση και τα όσα είχε πει και ο επικεφαλή ε, τη ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συμβουλίου τη Κοινοβουλευτική του Συμβουλίου τη Ευρώπη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα εσωτερικά. Πρόκειται για τροπολογίε τι οποίε ε, έχουμε υποβάλει ήδη γραπτό και μπορούμε να ομαδοποιήσουμε σε τρει κατηγορίε. Πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε τι τροπολογίε οι οποίε στόχο έχουν να προβάλλουν το έργο και τι προδιαγραφέ του Συμβουλίου τη Ευρώπη, ώστε αυτέ να αντικατοπτρίζονται, αυτά να αντικατοπτρίζονται σωστά, με ιδιαίτερη έμφαση στο ότι πρόκειται για την κορονίδα τη προστασία των σπουδών δικαιωμάτων σε επίπεδο Ευρώπη. Επίση, η δεύτερη κατηγορία των τροπολογιών μα. αναφέρεται στην, η στόχο έχει να προβάλλει τα, ε, τις δυνατότητες προσφυγής ε, που προβέλεπονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις διαδικασίες του, ιδιαίτερα για την ε, καταπολέμηση του εμπορίου εις βάρος γυναικών και παιδιών. Και ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε το ρόλο του συντονιστή διακίνηση γυναικών και παιδιών έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί και να μην λησμονηθεί ο ρόλο του υπό τη σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη κατά του ε, λαθρεμπορίου εις βάρος ανθρωπίνων όντων και ιδιαίτερα τον ε, υπογραμμίζουμε και το μηχανισμό συνεργασία που, που ε, προβλέπει αυτή η σύμβαση και που ήδη λειτουργεί. Επίση, προτείνουμε να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και κυρώσουν τη σύμβαση για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση ή καταχρήση. Ναι, ναι, θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε. Και ε, πάλι η επόμενη κατηγορία των τροπολογιών μας αναφέρεται στη μετανάσταση και το άσυλο και τελευταία μου γενική παρατήρηση θα ήθελα να υπογραμμίσω τις ανησυχίες μας ως προς την έμφαση που δίνεται για τις διαδικασίες της μετανάστευσης και του ασύλου στην, ε, στο κείμενο της Στοκχόλμης, χωρίς όμως να ε, μια ματιά ουσιαστική στον άνθρωπο, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους άνδρες που αναγκάζονται οι ίδιοι να... Λυπάμαι που σας παίρνω το λόγο κυρία. Λυπάμαι. Πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η κυρία Βαμικίενε από το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ και εσάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Εδώ και 20 χρόνια όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου δεν μπορούσαμε ίσως ακόμα να φανταστούμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προεδρεύεται από έναν πολιτικό της γεωγραφικής μας περιοχής. Πραγματικά κάτι τέτοιο το να συμβεί είναι ένα θαύμα ιδιαίτερα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δύο δεκαετίες διαδέχτηκαν εκατοντάδες χρόνια σκλαβάς και μιζέριας που χαρακτήριζαν ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Τώρα όμως συζητάμε θέματα πολύ πιο σημαντικά όπως το θέμα του προγράμματος της Στοκχόλμης. Εκτιμούμε θετικά το ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα μπορέσουμε να περάσουμε στην επαναξιολόγηση των εγκλημάτων τα οποία διέπραξαν και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Τα κοινοβούλια των κρατών μελών κάνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες αυτές και οικονομικά και πολιτικά φυσικά Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψεις σε διαφορετικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες κουβαλούν εντελώς διαφορετικές ιστορικές θα έλεγα εμπειρίες και αυτές ακριβώς οι εμπειρίες μερικές φορές οδηγούν τα κοινοβούλια στο να κρατήσουν διαφορετικέ θέσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ακριβώς το τι είχε συμβεί με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη και δεν μπορούμε παρά να είμαστε απόλυτα ενωμένοι στα πλαίσια του ολοκληρωτισμού. Οι μέθοδοι τις οποίες ακολούθησαν οι ολοκληρωτικοί ηγέτες στην Ευρώπη ήσαν ίδιες. Μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανισμοί, δολοφονίες. Και άλλα μέτρα καταστολής τα οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί για να σεβαστούμε από εδώ και πέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αντίληψη για όλα αυτά τα εγκλήματα του παρελθόντος. Επί τη βάση ακριβώς της σεβασμού της αρχής της, των αρχών της μη διάκρισης δεν μπορούμε να αποφύγουμε να κοιτάξουμε το ιστορικό μας παρελθόν. Εγώ είμαι υπεύθυνη και της ε, Λιθουανικής Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στον ΟΑΣΕ και πέρυσι υπήρξε μια δήλωση η οποία ξεκάθαρα ε, καταδίκασε τα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη. «325 ε, βουλευτές υπέγραψαν την δήλωση αυτή» και μόνο οκτώ μάλλον από αυτούς απέριψαν την πρόταση αυτή, μια πρόταση επαναλαμβάνω καταδίκη των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Συνεπώς έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα και νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε άλλωστε και ο κύριος Μετβέντεφ, ο οποίος καταδίκασε πλήρως τα σταλινικά εγκλήματα, ανοίγουν ένα νέο δρόμο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Παρακαλώ τους συναδέλφους, επαναλαμβάνει ο κύριος Μπούζεκ, να σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Ε, ε, ε, ο κύριος Κοέλιο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο λεπτά, τρία λεπτά, συγγνώμη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο συζητάμε σήμερα το απόγευμα, και που θα το συζητήσουμε και πιο ενδελεχώς ε, στις ομάδες εργασίας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Καθώς περνάμε από μια Ευρώπη που ήταν κοινή αγορά σε μια πραγματική Ευρώπη των πολιτών. Και όσοι είναι υπέρ μια τέτοια Ευρώπη χαίρονται που συζητάμε το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη. Υπάρχουν τρεις, ε, τρία πράγματα που πρέπει να τονίσουμε. Η πρώτη δοκιμασία είναι η δοκιμασία ευθύνη. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ότι αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Ε, πέρασε με καλό βαθμό αυτή η δοκιμασία. Όπως και όταν το Συμβούλιο συμφώνησε ε, κάποια θέματα να ρυθμιστούν και να ληφθούν υπό τη συναπόφαση πιο ταχαίως από άλλα ζητήματα. Ε, βέβαια υπήρχαν κατηγορίες ότι όταν το Συμβούλιο έπρεπε να ακούει το Κοινοβούλιο τα πράγματα καθυστερούν. Φυσικά όταν χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες της ομοφωνίας τα πράγματα κινούνται πολύ πιο αργά από ό,τι με την απόφαση. Υπάρχουν και άλλες δύο δοκιμασίες. Η δοκιμασία της συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα καθώς και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, στον τομέα της, ε, του ελέγχου της επικουρικότητα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ε, ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, το Εθνικό, και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Τώρα και η ΜΕΝ και η ΔΕ ε, θα έχουν περισσότερε εξουσίε. Υπάρχει και η δοκιμασία τη αποτελεσματικότητα. Δεν έχει νόημα να κάνουμε ωραίους λόγους στους πολίτες ε, της Ευρώπης για την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αλλά όταν πρόκειται να περάσουμε νομοθετήματα δεν κάνουμε τίποτα. Δεν τα καταφέρνουμε. Φυσικά υπάρχουν τομεί όπου πόρο απέχουμε από το να κατακτήσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα. Σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα, δεν τα πάμε πολύ καλά. Η δεύτερη γενιά του Σέγγεν θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ ήδη, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ όλοι αυτοί οι κανόνε δηλαδή και ενδεχομένω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα τεθούν σε ισχύ. Αυτό το σύστημα έχει καθυστερήσει. Και όσο καθυστερεί, δεν θα υπάρχει ένα σωστό σύστημα ευρωπαϊκών θεωρήσεων. Επίση, στον τομέα τη δικαιοσύνη θα έπρεπε να είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος ε, Δεκεμβρίου του 2009, αλλά δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Ε, καθώς και στο άσυλο και στη μετανάστευση. Και εκεί έχουμε καθυστερήσει για να, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των ε, στόχων. Έχουμε περάσει τη δοκιμασία της ε, υπευθυνότητα, αλλά έχουμε άλλες δύο δοκιμασίες, συνεργασία και αποτελεσματικότητα που ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Χωρίς αυτές τις δύο δοκιμασίες αποκλείεται να ολοκληρώσουμε την οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών η κυρία Καμίλ από το Βέλγιο, το Βελγικό Κοινοβούλιο. Monsieur Χιλιάδες άνθρωποι από τον Νότο ρισκάρουν τη ζωή τους κάθε χρόνο για να έρθουν στις χώρες μας, περνώντας από τα διάφορα στενά και θαλασσοπνιγόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν οι Βέλγοι σοσιαλιστές θεωρούμε ότι οι πολιτικές απαντήσεις της Ένωσης δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ικανοποιητικές. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα για μας είναι αυτή η οδηγία του Ιουνίου 2008, η οδηγία επαναποτρισμού. Εμείς καταδικάζουμε αυτήν τη δεξιάζουσα ιδέα ορισμένων κομμάτων που λένε ότι η μετανάστευση πρέπει να είναι στοχευμένη και προγραμματισμένη. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ως πρώτο, ως πρώτο δικαίωμα το να μπορεί κάποιος να αναπτυχθεί στην ίδια του τη χώρα αναπτύσσοντας σχέδια, προγράμματα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, στη χώρα του. Διότι καθένας δεν παίρνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση το δρόμο της εξορίας και των βασάνων. Βεβαίως, ανά τον κόσμο πάντα θα έχουμε, έστω και αν λύσουμε όλα τα οικονομικά προβλήματα, Πάντα θα έχουμε ανθρώπους που τους διώχνουν, ανθρώπους που τους φυλακίζουν, που τους εξορίζουν. Πρέπει λοιπόν εμείς να διαφυλάξουμε τις αρχές Πρέπει λοιπόν εμείς να διασφαλίσουμε τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη της Γενέβης. Θα πρέπει να διαφυλάξουμε όμως για όσους έρχονται εδώ τα κοινωνικά τους δικαιώματα για να μην υποσκάψουμε και τα δικαιώματα συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των ιδίων μας των κατοίκων. Πρέπει λοιπόν μεταξύ μεταναστών και ντόπιων ε, ηθαγενών τέλο πάντων εργαζομένων να υπάρχει ισονομία. Πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις αλλά και το δικαίωμα της ε, οικογενειακής επανένωσης. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να προασπίσουμε αυτές τις προοδευτικές ιδέες σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας. Ο Πολωνός συνάδελφος έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι η αφορμή της σημερινής μας συνεδρίασης. Στόχος του προγράμματος αυτού, του προγράμματος της Στοκχόλμης, είναι να προωθήσει την Ευρώπη στις τρεις βασικές, στον τομέα των ελευθεριών, στον τομέα της δικαιοσύνης και στον τομέα της ασφάλειας φυσικά βιώνουμε θα έλεγα τις συνέπειες σήμερα των αποφάσεων που οδήγησαν στην ελευθερία της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης την οποία γιορτάσαμε πριν από μία εβδομάδα. Ήταν καρπός μιας τεράστιας προσπάθειας της προσπάθειας για την απόκτηση της ελευθερίας η ελευθερία δεν ήταν ποτέ δεδομένη για κανέναν και οι προσπάθειες που έγιναν και στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη επιτέλους οδήγησαν σε αυτή. Νομίζω ότι οι ελευθερίες, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη είναι οι τρεις τομείς στους οποίους μπορούμε να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών. Ήδη η πρώτη συνάντηση στο Τάμπερε που έβαλε τα θεμέλια για τη συνεργασία μας στον τομέα αυτό έχει προσφέρει θετικά αποτελέσματα. Μαζί με τις αποφάσεις της Χάγης δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες να ζήσουν σε άλλα κράτη-μέλη, να ταξιδέψουν ελεύθερα σε άλλα κράτη-μέλη. Έτσι μόνο η Ευρώπη πραγματικά ενοποιείται και φτάνουμε ίσως σε μία περίοδο της ε, Ευρώπης της Αναγέννησης όπου οι Ευρωπαίοι, ιδιαίτερα οι νέοι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι σπουδαστές ε, θεωρούνται πολίτες του συνόλου της Ευρώπης, δεν είχαν συγκεκριμένη εθνική ιδιότητα. Θα πρέπει λοιπόν τις ανάγκες των πολιτών μας και τις ανάγκες των νέων πολιτών της Ευρώπης να τις καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο τομέας των ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης αφορά το σύνολο των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης και ακριβώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε στους τομείς αυτούς θα επιβάλλουν αν θέλετε και τον σεβασμό των Ευρωπαίων προς την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Αλλιώς ε, μια τέτοια προσπάθεια δεν θα στεφθεί από επιτυχία. Πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και μεταξύ των κρατών μελών για τη γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος της Στοκόλμης. Πολλέ φορέ δημιουργούνται ορισμένες αντιφατικές εικόνες σε σχέση με τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, σε σχέση με τις ελευθερίες και την ασφάλεια, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει την ζωή στην Ευρώπη. Απαιτείται λοιπόν συζήτηση και διαπραγμάτευση για να καλύψουμε τις ανάγκες και για ασφάλεια αλλά και για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και των ελευθεριών. Σα ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενο ομιλητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά ακούστηκαν σήμερα για κοινέ αξίε. Ένα κοινοβούλιο προφανώς περιλαμβάνει εντελώ διαφορετικές απόψεις, πολλές διαφορετικές απόψεις, όσες ακριβώ είναι και τα μέλη του και οι λαοί που το συναποτελούν θα έλεγα ε, ότι είναι πάρα πολύ θα έλεγα, αρνητικό το να θα λύσει κανείς να επιβάλλει κοινέ αξίες στο σύνολο των μελών ενός κοινοβουλίου και αυτό είναι κάτι που παραπέμπει σε συγκεντρωτικές μορφές διακυβέρνησης όπως είχε πει και ο Όργουελ ο οποίος θεωρούσε ότι ο έλεγχος του λόγου και ο έλεγχος της γλώσσας οδηγεί στον έλεγχο των μαζών και στον έλεγχο της σκέψης τελικά. Συνένεση πρέπει να υπάρξει. Μπορεί να προέλθει συνένεση από μια συζήτηση, εφόσον όμως η συζήτηση γίνεται με πραγματικός όρους ελευθερίας. Αλλά το να θελήσει κανείς να επιβάλλει όρους για τη συζήτηση, αυτό σημαίνει τέλος της ελευθερίας, αυτό σημαίνει τέλος της δημοκρατίας. Η βασική ελευθερία η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο ανώτατο θα έλεγα επίπεδο σεβασμού είναι η ελευθερία λόγου γιατί ε, φυσικά με περιορισμούς όπου υπάρχουν προσκλήσεις και προκλήσεις για διάπραξη βίας, για άσκηση βίας. Μόνο τότε μπορεί να ελεγχθεί η ελευθερία του λόγου. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο εκπρόσωπος του Κογκρέσου της Σουηδίας, ο κύριος Αλβάρο Κουέστο Μαρτίνες. Εγώ είμαι πρόεδρος Επιτροπής Δικαιοσύνης του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Να ξανασυστηθώ, το ξαναλέω. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τονίσω ότι με τη Λισαβόνα, την επικύρωση Λισαβόνας έχουμε μια τεράστια ευκαιρία μπροστά μας για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και ασφάλειας. οι πολίτες, άντρες και γυναίκες γίνονται πλέον το επίκεντρο όλης αυτής της προβληματικής. Υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα για να καταπολεμήσουμε την ίδια την οικονομική κρίση διότι αυτός ο χώρος είναι κάτι το θεμελιώδες και αποτελεί καταπέλκτη είναι ένα φρικτό νέο για την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, τις εργασίες της Κομισιόν θέλω να συγχαρώ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκτιμάμε πολύ θετικά πολλά από τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε τα ε, επόμενα ε, χρόνια. Είναι σημαντικότατες προτεραιότητες να επιμείνουμε ε, για το σχέδιο δράσης ε, του μέλλοντος. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην αμοιβαία ε, δικαστική αναγνώριση, ε, στην εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των εγγύσεων στις δικαστικές διαδικασίες. Θα πρέπει να αναπτύξουμε στοιχεία που βελτιώνουν την προστασία των θυμάτων. Δεν μπορούμε εμείς ε, τα θύματα να τα αποξενώνουμε από αυτόν τον χώρο της ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει και στη σύμβαση για, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν εμείς να προστατεύσουμε τα πιο ευαίσθητα άτομα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία μεταξύ των φίλων Θα πρέπει να προστατεύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα θύματα ε, κακοποίησεων. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις ευρωπαϊκές εισαγγελίες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην δικαστική συνεργασία σε θέματα ε, οικογενειακού και αστικού δικαίου. Ο χώρος ε, ελευθερίας ε, δικαιοσύνης και ασφάλειας είναι ένα καταπληκτικό νέο για τους Ευρωπαίους πολίτες και ένα φρικτό νέο για την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Ο λόγος δίδεται σε εκπρόσωπο του Συνδικού Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε κατά τρόπο αποτελεσματικό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας εν γέννη. Πολλά είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και βέβαια υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν μέσα από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Το κόμμα της αριστεράς ε, έχει ε, διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις, συμβάλλοντας έτσι ως προς την επιτυχία του προγράμματος της ε, Στοκχόλμης. Θα ήθελα λοιπόν να προσυπογράψω και εγώ τα όσα υπόθηκαν νωρίτερα από αρκετού συναδέλφου και ιδιαίτερα από την εκπρόσωπο του Βελγίου για τα θέματα του ασύλου και τη λαθρομετανάστευση. Πάνω απ' όλα θέλουμε να αναλυφθούν μέτρα τα οποία θα αποκλείουν τον, τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών. Και έχουμε από το Σπουδικό Κοινοβούλιο λάβει μέτρα νομοθετικά τα οποία απαγορεύουν την αγορά σε τέτοιου είδου σεξουαλικές υπηρεσίες. Όμως θα πρέπει όλοι να συμπράξουν. Αυτό προβλέπει άλλωστε το σουηδικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη καλύτερα. Ε, μιλούμε για την προστασία των ομοφιλοφίλων, αλλά και κάθε ατόμου από την σεξουαλική εκμετάλλευση και εξασφαλίζουμε με τις προτάσεις μας το δικαίωμα για την κάθε γυναίκα να ελέγχει και να έχει την απόλυτη ελευθερία στο σώμα της. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναλυφθούν τέτοιου είδους μέτρα και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. όπως επίσης και ε, να αναλυφθεί κάθε, το οποίο, μέτρο το οποίο θα σήμαινε ε, παρέμβαση στην ακαιρεότητα του ανθρώπου. Αυτά νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν μέτρα ουσιαστικά για την προστασία του καθενός, οποιαδήποτε επίσης. Θα ήθελα όμως πολύ να αναφερθώ και στο ζήτημα του ασύλου. Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις έτσι ώστε να μπορεί κανείς νόμιμα να ζητεί και να εξασφαλίζει το άσυλο έτσι ώστε να υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες και να μην είναι κανείς υποχρεωμένος να καταφεύγει ή να πέφτει στα χέρια των διακινητών και να μην κινδυνεύει να επαναπατριστεί της βίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο το Προεδρείο στον συνάδελφο τον Περ Βέστερμπεργκ Το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την τόσο σημαντική συνεδρίαση. Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι θέλουμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη ε, μέσα από τις ελπίδες των ε, πολιτών, ε, μέσα από τα ιδεώδη των, ε, της των ελευθεριών, της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι ωραία λόγια, ωραία διακόσμηση συνήθως στην ορολογία μας, στην κοινοβουλευτική, αλλά στην πράξη αποδεικνύονται μόνο ψημίθια και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις εξελίξει των τελευταίων δέκα ετών με, τις, ε, με τους πολυδατικούς ελέγχους στα σύνορα, με την αποτυχία στην, στον έλεγχο των ανατολικών σύνορων, όπου έχουμε ένα απόλυτα ε, ανοιχτό ε, πεδίο διακίνησης από την Ελλάδα στη Δανία μέσω της Φιλανδίας όπλων, ναρκωτικών, ανθρωπίνων όντων χωρίς κανένας να μπορεί να ελέγξει τα σύνορα τα ανατολικά της Ευρώπης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ολόκληρη οργάνωση, ένα σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο στηρίζεται σε πραγματικότητα διαφορετική ουσιαστικά από αυτήν την οποία συναντά στην καθημερινή του ζωή ο πολίτης, μέσα στην οποία ζει ο πολίτης. Και πρέπει, πλέον να δούμε την ε, μετανάστευση ως μέσα στις ε, πραγματικές της διαστάσεις και να αφήσουμε τα ωραία λόγια. Ε, ακούμε τις επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακούμε το δικαστήριο το οποίο ζητά να αλλάξουμε πολιτική, αλλά για να μιλήσω ανοιχτά, δεν μπορούμε να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ελεγγύη στην Ευρώπη, γιατί κανείς δεν ρωτάει το Δανό, το Γερμανό, το Γάλλο, πώς ζει και πώς μπορεί να συνεχίσει να ζει μέσα σε ένα χώρο ο οποίος έχει επεκταθεί τόσο που ε, να θεωρείται ότι μπορεί να χωρέσει κάθε δυνατή θρησκεία, ακόμη και το Ισλάμ, άκουσον άκουσον. Εδώ ακριβώς ε, ε, έχουμε τα προβλήματα και μετά μας μιλάτε για ρατσισμό. Όταν όμως ο πολίτης είναι δυσαρεστημένος, όταν βλέπει καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω αυτών των ε, φαινομένων, τότε δεν μπορείτε να τον κατηγορείτε για ρατσισμό, δεν μπορείτε να μιλάτε για ορολογία του μίσους. Πρέπει να πάρετε τον πολίτη στα σοβαρά υπόψη. Και χρειαζόμαστε μια Ευρώπη της ασφάλειας, μια Ευρώπη της δικαιοσύνης και πάνω απ' όλα πρέπει να βρείτε απαντήσεις για τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες, γιατί η κατάσταση είναι πονίδιστη. Ευχαριστώ από, το, από την γερουσία της Τσεχίας, παρακαλώ, η επόμενη ομιλήτρια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίδετε το λόγο, Πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι, είχα την ευκαιρία να πάρω μέρος σε πάρα πολλές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις και εδώ στις Βρυξέλλες μεταξύ άλλων. Οι περισσότερες από τις συναντήσεις αυτές αφορούσαν περισσότερο θεσμικά και συνταγματικά θέματα Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη λοιπόν γιατί σήμερα δεν συζητάμε τέτοιου είδους θεσμικά και συνταγματικά θέματα αλλά ασχολούμεθα με θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και των δημοσίων ελευθεριών. Ευτυχώς και ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία επικύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες μέλη για την ε, υποστήριξη την οποία έδωσαν στη δική μου χώρα, στην Δημοκρατία της Τσεχίας, ώσπου να επικυρώσει τη συνθήκη. Εμείς η πολιτική μου δύναμη, ο πολιτικός μου χώρος έδωσε σκληρές μάχες για να μπορέσουμε να επικυρώσουμε τη συνθήκη ακριβώς επειδή ε, συγκεντρώσαμε την προσοχή μας στα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην καρδιά των συμπολιτών μας. Και η ασφάλεια και η δικαιοσύνη φυσικά είναι τομεί οι οποίοι στην καθημερινότητά τους άπτονται της ζωής των πολιτών της χώρας μου και όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Προφανώς η διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα θα είναι μια διαδικασία γεμάτη εμπόδια και καθυστερήσεις. Θα υπάρξουν ίσως διαφορετικές ερμηνείες στα διάφορα κράτη-μέλη για τα ίδια κείμενα και μπορούμε να προσπαθήσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα αυτά και σε επίπεδο διακοινοβουλευτικών ε, συναντήσεων ή και σε επίπεδο της ΚΟΖΑΚ η οποία ξέρετε ότι είναι μια διάσκεψη εθνικών κοινοβουλίων η οποία λειτουργεί συνεχώς άνω των 20 ετών και νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τη σωστή της λειτουργία. Συνεπώς πέραν της ΚΟΖΑΚ θα πρέπει να ξεκινήσει ε, μια συζήτηση η οποία να έχει σαν στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και, του νέων, και των νέων μορφών εθνικισμού που αναθείονται σε διάφορες χώρες και δημιουργούν ανησυχίες. Υπάρχουν προβλήματα επίσης όπως της ανακύκλωσης του βρώμικου χρήματος, του οργανωμένου εγκλήματος, του εμπορίου ή λαθρεμπορίου ναρκωτικών Όλα αυτά είναι πολλά προβλήματα τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα μπροστά μας. Μόνο αν τα λύσουμε θα προσφέρουμε μια ασφαλή Ευρώπη στους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο τώρα ο κύριος Γκουτιέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είχε πολλά πλεονεκτήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι βέβαιο, τουλάχιστον για την Ισπανία. Βέβαια δημιούργησε και ορισμένα ζητήματα. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης οδήγησε σε ένα έλλειμμα ασφάλειας. Διότι εμείς καταργήσαμε τα σύνορα για τους εγκληματίες και σε μεγάλο βαθμό διατηρήσαμε τα σύνορα για τους αστυνομικούς και τους δικαστές. Εγώ πιστεύω από τη διαδικασία του Τάμπερε πριν από 10 χρόνια έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο να γκρεμίσουμε αυτά τα σύνορα για τους αστυνομικούς και τους δικαστές. Όμως παραμένει ακόμα πολλής δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως όσον αφορά στην νομική συνεργασία. Οι, οι αστυνομικοί ανταλλάσσουν με μια σχετική ευκολία τις ε, πληροφορίες τους, αλλά όταν χρειάζεται μια συγκεκριμένη ανταλλαγή πληροφοριών συνεργασία πάνω σε μια ποινική υπόθεση, η ροή των πληροφοριών δυσκολεύει. Πρέπει να εγγυθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Σε μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αμφισβητήσουν την νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαντήσει σε προκλήσεις όπως είναι η ασφάλεια και η καταπολέμηση του, οργανωμένου εγκλήματος. Λοιπόν, εγώ θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στην ατζέντα της Στοκχόλμης αλλά κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Όχι να λέμε ότι απλώς εμείς ε, θα διευρύνουμε την ατζέντα αυτή. Όχι, πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί πάνω στα θέματα τα οποία μας θέτει το ίδιο το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Πρέπει λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια να είναι πολύ απαιτητικά προς τις κυβερνήσεις για να μπορούμε να έχουμε προγράμματα που θα εγγυώνται αποτελεσματικά την ασφάλεια των πολιτών τους που αποτελούν και την πρώτη ανησυχία σήμερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τερέσα Χιμένες Μπεσερίλ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, señor presidente. Ε, εγώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένας καλύτερος, ένα καλύτερο μέρος από ότι εδώ για να μιλήσουμε για τα θύματα της τρομοκρατίας. Εμείς ε, μιλάμε εδώ για το πρόγραμμα της Στοχόλμης ε, που αφορά στην ασφάλεια, στην ελευθερία και στη δικαιοσύνη. Αυτά είναι και τα τρία πράγματα που ζητούν τα θύματα της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ασφάλεια, δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη. Το είπε και ο κύριος Κοέγιο προηγουμένως. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Εγώ το λίγο καιρό που έχω σε αυτό το κοινοβούλιο διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα σχετικός φόβος για την τρομοκρατία. Μιλάμε σχετικά λίγο για την τρομοκρατία. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και υποφέρουμε από αυτό. Το υποφέρει τώρα η χώρα μου η Ισπανία αλλά τα τράβηξε και η Ιταλία και η Ιρλανδία και πολλές άλλες χώρες στο παρελθόν και όλοι είμαστε εν θύματα της τρομοκρατίας. Εγώ ε, είμαι σε θέση να μιλήσω γι' αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς ε, να φοβόμαστε να μιλάμε για την τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει εμείς να σιωπάμε γύρω από τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας θεωρώντας ότι όταν εμείς προωθούμε τις διεκδικήσεις των θυμάτων μειώνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ δεν θέλω εδώ να μιλάμε ούτε για δικαίωμα των θυμάτων, ούτε για τα δικαιώματα των τρομοκρατών. Θέλουμε να μιλάμε για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Ζητώ αλληλεγγύη από τα 27 από όλε τι 27 χώρε τη Ένωση, ούτω ώστε και να βοηθήσουν την Ισπανία και τα θύματα της τρομοκρατία, προασπίζοντα τα αιτήματά τους. Θα έπρεπε λοιπόν εμεί να προχωρήσουμε σε μία εναρμόνιση της νομοθεσίας τώρα με τη Λισαβόνα για την προστασία των θυμάτων και τους νόμους που προστατεύουν τα θύματα. Να καταφέρουμε να έχουμε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας και μέσα από το πρόγραμμα της Στοκόλμης νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητέ. Θα κλείσω γι' αυτό το λόγο τον κατάλογο των ομιλητών. Ούτω ώστε μετά τι 5 ώρα το απόγευμα να πάμε στι ομάδε εργασία. Και μάλιστα θα μειώσω και το χρόνο για κάθε παρέμβαση. Δύο ε, λεπτά το κάθε άτομο. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι απαραίτητο αν θέλετε να μιλήσουν όλοι που είναι γεγραμμένοι στον κατάλογο μιλητών. Σκίδη Κουκούμα από την Κυπριακή Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, η δημοσίευση από τη Σουηδική Προεδρία του προσχεδίου του προγράμματος της Στοκόλμης για την περίοδο 2010-2014 μας θέτει και πάλι ενώπιον των ζητήματος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη τις ατομικές και δημοκρατικές ελευθερίες. οφείλω εξ αρχής να καταθέσω τις θέσεις μου για μια σειρά πολιτικών που ακολουθεί η ευρωπαϊκή ένωση και που προβλέπεται να επεκταθούν μέσα από το προτινόμενο πολιετές πλαίσιο πολιτικής στα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. η συνεχής ενίσχυση των κατασταλτικών θεσμών και πολιτικών δεν είναι η απάντηση στα θέματα ασφάλειας και δικαιοσύνης. θέτω το θέμα της ευρωαστυνομίας ένα σώμα καθολική αστυνόμευση των κοινωνιών το οποίο δεν υπόκειται σε ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο και ταυτόχρονα διαθέτει εξουσίες που φτάνουν μέχρι την παρακολούθηση όχι μόνο των αποδεδειγμένων εγκληματιών αλλά και υπόπτων ή ακόμα και των λεγόμενων πιθανών εγκληματιών. οι πρακτικές συλλογής προσωπικών δεδομένων βιομετρικά στοιχεία δαχτυλικά αποτυπώματα γενετικών υλικών το οποίο η θεσμοθέτηση ολοκληρώνεται με τη συμφωνία σέγγεν δεύτερη γενιά και τη συνθήκη προύμ αποτελούν ευθυγράμμιση με όσα ακριβώς εφαρμόζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική μετά την πτώση των δίδυμων πύργων το 2001 και υπό το πρόσχημα πάταξη της τρομοκρατίας εισβάλλει θεσμοθετημένα πλέον σε θέματα πολιτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και χτυμένα που οι λαοί κέρδισαν μέσα από διεκδικήσεις και αγώνες ξαφνικά απεμπολούνται στο όνομα πάταξης ενός εχθρού που εμείς ήδη δεν τον έχουμε καθορίσει όλα αυτά θέτουν σε συναγερμό κάθε υπερασπιστή των πολιτικών ελευθεριών. υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας συρρυκνώνεται η ελευθερία έκφρασης και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής τη στιγμή μάλιστα που οι αντιλήψεις για την τρομοκρατία διαφέρουν ουσιαστικά δηλαδή τι περιλαμβάνεται τελικά στον όρο ριζοσπαστικοποίηση την οποία σπέβδει να προλάβει και να καταστήλει η ευρωπαϊκή ένωση όσοι δηλαδή εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνέργησαν στο αιματοκύλισμα τη γιουγκοσλαβίας και του ιράκ μπορούν να μα υποδείξουν τα όρια τη ελευθερία και τη ασφάλεια, αυτοί που ακόμα δεν μπορούν να αιτιολογήσουν τι πράξει του, όχι μόνο ηθικά αλλά ούτε καν βάση του διεθνού δικαίου; απολογούμε που πρέπει να σταματήσω. προετοιμάστηκα για τρία λεπτά αφού έχετε αλλάξει το χρόνο θα το σεβαστώ από την Τσεχική Γερουσία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την προσπάθειά σας, για την προσπάθεια της Προεδρίας σας, λαμβάνοντας υπόψη την τελική φάση της διαδικασίας κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω που σεβαστήκατε και τα συνταγματικά δικαιώματα των κρατών μελών. Νομίζω ότι, είναι, ότι κρατήσατε την καλύτερη στάση που μπορούσατε να είχατε κρατήσει και αυτά είναι θαυμάσια νέα για του Ευρωπαίου πολίτε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Μπούζεκ που οργάνωσε αυτή τη συνάντηση και που έγινε και να τον συγχαρώ που έγινε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι μικρό αυτό το κατόρθωμα. Η απόφαση της τσεχικής ε, γερουσίας για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα συζητηθεί αύριο από τον συνάδελφό μας, τον κύριο Γκρούλιχ. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για μια πρόταση, για μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου στο σημείο 13 μιλάει ε, για τον έλεγχο της Europol, Eurojust και Frontex. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται και στον έλεγχο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι κάτι το οποίο μας το υποσχέθηκε η Γαλλική Προεδρία στην Πράγα και είμαι σίγουρος ότι θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνάντηση της ΚΟΖΑΚ. είναι κάτι το οποίο παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ στα εθνικά κοινοβούλια εδώ και καιρό. Ε, θα ήταν ατυχέ να γίνει ο έλεγχο μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου, μην, ξέρετε, μην ξεχνάτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πολλή εμπειρία σε αυτά τα θέματα, ενώ τα εθνικά κοινοβούλια έχουν αντίθετα. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί σα σε αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα περιμένουμε το βασικό έγγραφο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω μα υποσχέθηκε, το οποίο εν συνεχεία θα συζητήσουμε στην ΚΟΖΑΚ και με μονόμενα τα εθνικά ε, κοινοβούλια, αλλά στην Κόζακ θα τα συζητήσουμε μεταξύ μα και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο εργασία. Σα ευχαριστώ. Χέιτι Χάουταλα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε τον λόγο. Εγώ εδώ θα μιλήσω ως αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλω να σταθώ στην εξωτερική διάσταση του προγράμματος της, λισαβόρ ε, Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για την εξωτερική διάσταση διότι οι διάφορες αυταρχικές εξωτερικές δυνάμεις μας ξεμπροστιάζουν κάθε φορά που ξέρουν δηλαδή ότι εμείς έχουμε την πρωτοπορία σε αυτό τον τομέα και κάθε φορά που στα διεθνή φόρα εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία μας ξεμπροστιάζουν λέγοντας ότι εσείς είστε διαφορετικοί και ξέρουμε πάρα πολλές φορές ότι όταν ενεργούμε σε μεμονωμένο επίπεδο στα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη κοιτάζουν να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο, ακριβώς για να μην εκτίθενται σε αυτές τις κριτικές. Το δικό μου το κοινοβούλιο, το Φιλανδικό Κοινοβούλιο, θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα και αυτό λόγω της εξωτερικής διάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ λοιπόν από τα Εθνικά Κοινοβούλια να τονίσουν το πόσο σημαντική είναι αυτή η εξωτερική διάσταση του προγράμματος της Στοκχόλμη. Πολύ σημαντικό για το διεθνές δίκαιο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν και τη λιδία λίθο των εξωτερικών μας σχέσεων. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε όσο το δυνατόν πιο τονισμένη αυτή την εξωτερική διάσταση και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα τεράστιο έργο μπροστά μας. Αν θέλουμε να αποφύγουμε η Επιτροπή να τελειώνει τις εργασίες νερώνοντας όλη την προσπάθεια. Ε, Κύριος Κάπλαν, από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω στους πολίτες και στους βουλευτές το ερώτημα ε, τι Ευρώπη θα χτίσουμε με αυτό το πρόγραμμα. Όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Χάρτα θα είναι υποχρεωτική νομικά για όλα τα κράτη-μέλη. Και αντί για την Ευρώπη των πολιτών, που είναι ο τίτλος της σημερινής μας συζήτησης, ίσως θα πρέπει να χτίσουμε μια Ευρώπη ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε σε επίπεδα ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας που είναι ο κωδικός, ε, τα μαγικά λόγια ε, σε αυτά τα κείμενα για όλους τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έγγραφο που μιλάει για τα δικαιώματα και τη χάρτα ε, σε εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες ε, παραδείγματος χάρη κά, κάποιες βορειοαφρικανικές χώρες όπου παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αφαιρούν το νομικό καθεστώς κάποιων ανθρώπων. Ε, επίσης υπάρχει πρόβλημα για τους απάτριδες ανθρώπους. Ε, όλα αυτά με ανησυχούν πάρα πολύ. Το κείμενο αυτό ε, νομιμοποιεί όλους τους αυτούς τους ανθρώπους. Η Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ελπίζω να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Είναι μια δοκιμασία για τη συνείδησή μας. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να μην επαναλάβουμε, πέντε χρόνια, να μην επαναλάβουμε κάποια, κάποιες απόψεις ε, ε ανησυχητικές που ακούσαμε ακόμα και σήμερα. Ε, και ελπίζω στα κείμενά μας να μην να υπάρξουν στοιχεία Ισλαμοφοβίας κτλ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλιτς από το Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Πολωνικής Βουλής. Το 2004 ήμουν υπουργό Εσωτερικών στην Πολωνική Κυβέρνηση και παρακολούθησα από πάρα πολύ στενά την προπαρασκευαστική περίοδο του προγράμματος της Χάγης και παλιότερα του προγράμματος του Τάμπερ. Απευθύνω λοιπόν μια έκκληση προς τον πρόεδρο Μπούζεκ έτσι ώστε να μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο και το ταχύτερο δυνατόν οι προβλέψεις τις οποίες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Χάγης να αναλυθούν σωστά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε σε κάποια στιγμή να εφαρμοστούν. Πάρα πολλά σημεία του προγράμματος της Χάγης δεν έχουν καν μεταφραστεί ουσιαστικά στις ε, γλώσσες της Ένωσης. Ένα δεύτερο θέμα. Πριν μάλλον περάσω στο δεύτερο θέμα θα ήθελα φυσικά να συγχαρώ προσωπικά τον πρόεδρο και εξ ονόματος της πολωνικής ε, αντιπροσωπείας. Πρώτη φορά μπορώ και το κάνω αυτό δημόσια για την θέση την οποία ανέλαβε. Σχετικά με τις θέσεις τώρα τις οποίες έχει ήδη παρουσιάσει η Σουηδική Προεδρία θα ήθελα να διαπιστώσω μία κάποια μικρή αντίφαση θα έλεγα ανάμεσα στα μέτρα υπέρ των δημοσίων ελευθεριών και από την άλλη στις ανάγκες για την ασφάλεια των πολιτών, για την άμυνα των πολιτών. Έχω, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνεργασία ανάμεσα στις δυνάμεις της αστυνομικές και τις δυνάμεις καταστολής από τη μία και από την άλλη ε, τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές εμπειριών και χρηστών πρακτικών στα πλαίσια της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση όταν προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του πολίτη να παραβιάζουμε τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τζορέγια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Yo creo que todos estamos de acuerdo en dos cosas que son importantes. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε γύρω από δύο πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Από τον Ιανουάριο και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετεί και αποφασίζει μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εσείς τα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε τη δυνατότητα να επαληθεύετε αν οι κανονισμοί και οι νόμοι που θα ψηφίζουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης παραβιάζουν ή όχι το δικό σα ουσιαστικό δίκαιο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν εκτός πια από αυτούς που δεν θέλουν καθόλου την Ευρώπη υπάρχει λοιπόν έλεγα σύμπτωση ότι πρέπει να ενοποιήσουμε, να προχωρήσουμε σε μια ομολογοποίηση του δικαστικού μας συστήματος και του ποινικού μας συστήματος. Θέλω να σας προειδοποιήσω με όλη την ειλικρίνη αγαπητοί συνάδελφοι ότι διατρέχουμε έναν κίνδυνο να μην λειτουργήσει όλη η διαδικασία. Ότι να γίνει τόσο πολύπλοκη η λειτουργία της Ευρώπης με την συνθήκη της Λισαβόνας, ούτως ώστε δεν είναι ένα βήμα προς τα μπρος, να είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Θέλω λοιπόν να σας προειδοποιήσω με όλη την ειλικρίνεια, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει ένα ρίσκο ως προς την ε, υπερκυριαρχική ή ριζοσπαστική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί από τα εθνικά κοινοβούλια διότι υπάρχουν πολλά ρεύματα στην σημερινή Ευρώπη τα οποία θεωρούν ότι τα κράτη, τα έθνη δεν θα πρέπει να απαρνηθούν τίποτα. Άμα δεν είχαμε όμως απαρνηθεί το φράγκο, το, το, μάρκο, τη λιρέτα δεν θα είχαμε ευρώ. Χρειάζεται λοιπόν να σταματήσουμε αυτήν την άκαμπτη κυριαρχίστικη ε, ερμηνεία του ποινικού δικαίου από τα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, στο πρόγραμμα της Ευρώπης. Ο Λόρδος Μπόουνες ε, από την Βουλή των Λόρδων Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε και μέλη των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Ευχαριστώ και τη Σουηδική Προεδρία για την προσπάθεια την οποία έχει ήδη κάνει στα πλαίσια του προγράμματος τη Στοκχόλμης. Συμμερίζομαι την άποψη ότι έχουμε κοινέ αξίε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι προ συζήτηση. Το θέμα είναι πώ θα τι εφαρμόσουμε και πώ θα βοηθήσουμε έτσι ώστε να μην παραμείνουν απλέ ιδέε. Το πρόγραμμα τη Στοκχόλμης έτσι όπω έχει διατυπωθεί, κύριε Πρόεδρε, είναι ιδιαίτερο φιλόδοξο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στο εσωτερικό στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς και η αντίστοιχη Επιτροπή της Ανοβουλής. Αλλά αν πρέπει να πετύχουμε ορισμένους στόχους και θέλουμε να τους πετύχουμε, πρέπει να κατορθώσουμε ορισμένες προτεραιότητες. Δεν θα πετύχουμε τα πάντα μέσα σε μια πενταετία και ακριβώς εφόσον δεν πετύχουμε να περάσουμε τις προτεραιότητές μας, τότε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρήσουν ότι το πρόγραμμα της Στοχόλμης δεν είναι κάτι το σοβαρό για αυτούς. Πιστεύουμε ότι κάθε μορφή νέας νομοθετικής δουλειάς θα πρέπει να έχει διατυπωθεί σωστά, να έχει ελεγχθεί από τους πολίτες, να έχει ελεγχθεί από τους επαΐοντες και να έχει κριθεί από αυτούς σαν χρήσιμα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαν παράδειγμα, τα δικαιώματα των πολιτών στις δικαστικές διαδικασίες. Όταν ένας πολίτης δικάζεται σε μια χώρα με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετική γλώσσα, ε, και εκεί προφανώς πρέπει να γίνει κάτι και γι' αυτό ακριβώς η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών διαδικασιών και ποινών είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο από το να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε μεμονωμένα νομοθετικά θέματα στο σύνολο των 27 χωρών. Κοινέ πρακτικές έχουν νόημα μόνο εφόσον διευκολύνουν την επίλυση των διαφορών διακρατικά θα έλεγα, διαμεθοριακά, εφόσον βέβαια σεβόμεθα την αρχή της επικουρικότητας για να μην υπάρχουν ε, συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές νομικές δικαιοδοσίες. Ευχαριστώ Αλμπέρτο Μαριτάτη από την Ιταλική Γερουσία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε δύο λεπτά θα μπούσα απλώς να παριθμίσω τηλεγραφικά κάποιες έννοιες. Έτσι θα μιλήσω λοιπόν τρομερά λακωνικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι έφτασε η ώρα όπου η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να κάνει βαθιές αναλύσεις. Τις αναλύσεις τις κάναμε. Ε, όπως σωστά είπε και ο συνάδελφος ε, από την Ισπανία, έχουν πέσει τα σύνορα, κάτι που είναι θετικό, αλλά έπεσαν μόνο για τους εγκληματίες. Αλλά για τους πολίτες, ε, για τους ε, πολίτες όχι, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για τους ε, δικαστές, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν φραγμούς που θα πρέπει να απαλληφθούν. δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε τι κάνει το οργανωμένο έγκλημα με τόση ελευθερία. Ε, ο, η τρομοκρατία είναι πάρα πολύ δεδομένη, πάρα πολύ ελεύθερη. Θα πρέπει να υπάρξει μια κατασταλτική διεθνής απάντηση μέσω της δικαιοσύνης, μέσω κάποιων εργαλείων που έχουν ήδη κυρωθεί, όπως παραδείγματο χάρη οι κοινέ αστυνομικές ομάδες ε, σε πολλές χώρες, ε, μεταξύ των οποίων και η χώρα μου, όμως δεν έχουν επικυρώσει αυτά τα όργανα, ήδη από το 2002. Και η προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία ανήκα, ούτε η σημερινή έχει κυρώσει αυτό το μέτρο, ούτε η προηγούμενη στην οποία ανήκα. Θα πρέπει λοιπόν ε, το στομότερο δυνατόν να έχουμε εργαλεία πολύ χρήσιμα όπως το Europol και Eurojust. Χρήσιμα τι σημαίνει. Σε νομοθετικό επίπεδο να καθορίσουμε την δομή του, τι αρμοδιότητά του και προσοχή, συνάδελφοι, τι αρμοδιότητέ του. Γιατί αν του δώσουμε, όπω πρέπει να του δώσουμε, περισσότερε εξουσίε, περισσότερε δυνατότητε για να συντονίσουν, για να απαντήσουν με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο στο οργανωμένο έγκλημα, αυτέ οι υπηρεσίε, αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν και κάποιε ευθύνε ε, και η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει ανεύθυνη για αυτούς τους ε, οργανισμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε μια κάποια επίσης δικαστική συνεργασία. Τη χρειαζόμαστε πάρα αυτά. Χωρίς αυτό το στοιχείο δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν ούτε καν τα εθνικά συστήματα. Φανταστείτε πολλό δε μάλλον, ας πούμε, το ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ. Η Ελέν Φλότχα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει. Καταρχά, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι ύστερα από την κύρωση τη συνθήκη Λισαβόνα ε, τα νομοθετικά μα όργανα έχουν προ τώρα εξουσίε αξιολόγηση των πολιτικών ω προ την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνη εσωτερικών και ασφάλεια. Και δυστυχώ σημειώνω ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη ω προ ορισμένε έννοιε που θα έπρεπε να συζητηθούν περισσότερο σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Εμεί την ε, συνοδεία συνεδρία αυτή την ε, αποκαλούμε ευκαιρία για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των πολιτών. Γιατί υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, κίνδυνοι και παγίδε, δηλαδή ότι στο, ε, στην επικράτεια τη Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή επικράτεια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, δεν είναι ηθαγενεί δηλαδή ενό των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όμω ε, είναι υποκείμενα δικαίου, μάλιστα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, τα κράτη μας εξάλλου ε, αύριο μεθαύριο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρώνοντας ε, την κάρτα των δικαιωμάτων θα είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν τα δικαιώματα αυτά και να τα κάνουν σεβαστά. Γι' αυτό λοιπόν όταν έχουμε δικαιώματα ε, ε, τα οποία δεν γίνονται σεβαστά έχουμε πρόβλημα και βλέπω ότι είναι πολύ συσταλτική η ερμηνεία των θεμάτων της ε, ασφάλειας γιατί πιστεύω ότι θα έπρεπε να τη συζητήσουμε υπό την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας όπως ακριβώς την έχουν αναπτύξει τα Ηνωμένα Έθνη ο ίδιος ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έχει δώσει ορισμό της ανθρώπινης ασφάλειας και έτσι δίνει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα και προοπτικές για την Ευρώπη την ίδια. Βλέπω λοιπόν ότι λείπουν από αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης οι αναφορές στις διεθνείς δεσμεύσεις προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να μιλήσω με λόγια απλά, βλέπω ότι υπάρχει τεκμηρίωση και μέσω των οργάνων της, των, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, των Οργανώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Υπηρεσίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας θα πρέπει να εξάρουμε το έργο, αλλά οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τα ίδια τα κράτη-μέλη επίσης έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα και θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των προσπαθειών μα Η Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε πρέπει να εδράζεται πάνω σε αυτά τα θεμελιώδεις αξίες και πρέπει σαν στόχο να έχει να αποκαταστήσει αυτό το τεράστιο χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων και της πραγματικότητας όπω στην ε, υλοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Στέφαν Τσέναχ από την Αυστριακή Bundestag. Πρόεδρε ευχαριστώ και ζητώ απευθεία συγγνώμη από την Σουηδική Πρόεδρε, τους, τον Προεδρεύοντο, ε, ε, γιατί πολύ σύντομα θα αναφερθώ στα θετικά στοιχεία, το ζήτημα τη ελεύθερη κυκλοφορία των δικαιωμάτων κτλ. για να επικεντρωθώ στα αρνητικά. Φιλόδοξο λοιπόν το σχέδιο τη Στοκχόλμη, ναι, όντω, ε, πολύ καλά σχέδια, πολύ ωραία λόγια λέει ναι, αλλά και έχει πολλές αντιφάσεις, εμπεριέχει πολλές αντιφάσεις και βλέπω μεγάλη, ε, μεγάλο χάσμα μεταξύ των όσων ε, προβλέπονται να υλοποιηθούν και των δυνατοτήτων υλοποίηση αυτών. Πρέπει πιστεύω στα συμπεράσματα να σημειωθούν κάποια σοβαρά προβλήματα ως προς την αναδιάρθρωση, ως προς τους στόχους μας και, την, ε, και τον προγραμματισμό μας. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ σε κάποια ουσιαστικά ζητήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη που είναι κάποιε από τις βασικές αρχές του προγράμματο τη Στοκχόλμη, θα λέγαμε ότι έχει την πατρότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει και να λησμονήσουμε τους, ε, τη, σχέση αιτία και αιτιετού, την αναλογικότητα και πάνω απ' όλα τον έλεγχο που βλέπουμε να απουσιάζει από αυτό το πρόγραμμα, μέσα από αυτό το σύστημα ενημέρωση, δεν υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Και επίση, πριν από ένα χρόνο ακόμα συζητούσαμε τα θέματα τη μετανάστευση. Κατασκευάσουμε όμω ταυτόχρονα νέου στίχου για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης για να έχουμε υποτίθεται κάλυψη των ε, συνόρων μα, ενώ χωρί να έχουν ουσιαστικά εφαρμοστεί τα όσα είχαμε συμφωνήσει, προτείνονται νέε λύσει. Η αξιολόγηση του κινδύνου, όπω προτείνεται μέσα από το σύστημα για τη θεώρηση των διαβατηρίων, ουσιαστικά ανατρέπει το τεκμήριο τη αθωότητα. Και επίση θα ήθελα να αναφερθώ κατεπηγόντω ε, προ τη Σουδική Προεδρία και να τη στήσω να αναλάβει ε, δραστηριότητα ω προ το φαινόμενο τη ε, κυκλική μετανάστευση. Δεν υπάρχει προγραμματισμό και σχέδιο στα όσα μα προτείνεται εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταπάνη Τάλι από την Φινλανδία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πρόταση, το σχέδιο αυτού του πολιετούς προγράμματος αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στα ε, όσα είχε προτείνει και η φιλανδική κυβέρνηση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι συμπληρωματικό του προγράμματος του Τάμπερε και μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για την υλοποίηση της, ε, των ελευθεριών των πολιτών. Φυσικά πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετές διαφορετικές πτυχές στην υπόθεση αυτή και προκειμένου θα ήθελα να συγχαρώ την Σουηδική Προεδρία για το εξαίρετο έργο που έχει προσφέρει στην υπόθεση αυτή. Θα πρέπει όμω να είμαστε κάπω πιο συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα που θα έχουν λειτουργικά ε, θα μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη και θα δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να μην περιοριστούμε δηλαδή μόνο στα ευχολόγια. Θα θέλαμε να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα μέσα στο πρόγραμμα. Το δε σημαντικότερο εδώ είναι να εξασφαλιστούν αποτελέσματα. Μια αποτελεσματική δηλαδή ε, ένας αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων και μια ουσιαστική και αποτελεσματική διαδικασία για το άσυλο. Αυτά ήδη τα προετοίμασε με το έργο της και η Γαλλική Προεδρία πέρυσι ε, στο, στο προηγούμενο εξάμεινο και έτσι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια κοινή πολιτική ασύλου για το 2012. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα θέλαμε να δώσουμε στο γεγονό ότι πρέπει τα κράτη-μέλη τα κράτη -μέλη να αναπτύξουν μια κοινή πολιτική ασύλου. Είναι ανάγκη να έχουμε μια κοινή πολιτική ασύλου. Διότι μέχρι στιγμής είναι πολλές οι διαφορετικές ε, νομοθεσίες στα κράτη-μέλη οι οποίες δεν βοηθούν καθόλου στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κοινή νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Γκέραλτ Χέφνερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια και δεν έχω χρόνο Πρόεδρε, θα ήθελα πολύ σύντομα να περάσω στην ουσία στο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί δεν έχουμε πολλέ φορέ την ευκαιρία να συναντούμε εδώ συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητούμε σε αυτή την ευτυχή συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα, επί παραδείγματι. Και πρέπει να πω ότι εδώ εμεί είμαστε φορεί τη τεράστια ευθύνη με την οποία μα έχουν επιφορτήσει οι πολίτε τη Ευρώπη να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην πτυχή ποινικό δίκαιο, ε, τρομοκρατία δίκαιο σχετικό με την ασφάλεια και την ε, δικαιοσύνη. Εδώ βλέπουμε μόνο τέσσερις γραμμές μέσα στο πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης και θα ήθελα να σημειώσω ότι πέραν της μεγάλης χαράς που μας γεννά σε όλους το γεγονός ότι πριν από 20 χρόνια ε, τερματίστηκε η διχοτόμηση της Ευρώπης και μπορέσαμε να επανενωθούμε, να είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη και πάλι, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε ακόμη περισσότερες προσπάθειες, ακόμη περισσότερο μόχθο να καταβάλουμε για τους πολίτες αυτής της επανενωμένης Ευρώπης. Χρειάζεται να κάνουμε ακόμη πιο αλματώδη βήματα για αυτή την Ευρώπη, για να μην είναι μια Ευρώπη των ελίτ, αλλά μια Ευρώπη των λαών, για να έχουμε μια πραγματική Ευρώπη των πολιτών. Και εδώ ακριβώς το, European Citizens Initiative αποτελεί ένα σημείο εκκίνησης η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών μπορεί να αποτελέσει δηλαδή μια βάση που θα αποδειχθεί σε προσεχείς εβδομάδες και μήνες εάν όντως θα αποτελέσει ουσιαστική βάση ή αν τελικά θα λησμονηθεί. Εμείς πάντως ενθαρρύνουμε να ενταχθεί μέσα στον πολιτικό μας σχεδιασμό και θα θέλω να αφαιρθώ όχι μόνο στη συνεργασία των θεσμικών οργάνων, των θεσμών δηλαδή, αλλά και στις δυνατότητες που πρέπει να προσφερθούν στους πολίτες της Ευρώπης να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους, να έρχονται πιο κοντά σε δεν έχουν και την αίσθηση ότι και εμείς είμαστε κοντά τους, ότι μπορούν δηλαδή να συνδιαμορφώσουν την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θανάσης Παφίλης από την Ελληνική Βουλή. Αποτελεί πρώτα-πρώτα ηρωνία αυτό που υπόθηκε ότι προχωρούμε στην Ευρώπη των πολιτών. Και σας ρωτάω όλους αν ε, θεωρείτε ότι πάμε στην Ευρώπη των πολιτών γιατί για ένα τεράστιο θέμα που αφορά τη συνταγματική συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας, δεν τολμήσατε να κάνετε δημοψηφίσματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί όπου έγιναν οι Ελλάδα απάντησαν όχι και την Ιρλανδία με εκβιασμό και τρομοκρατία την σύρατε σε ένα ναι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε Ευρώπη των πολιτών, αλλά Ευρώπη των πολιεθνικών. Δεύτερο σχόλιο σε ό,τι αφορά το χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, Είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που διακήρυσε. Προωθείται ένα πρωτοφανέ αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο και κατασταλτικοί μηχανισμοί. Ο πιο αναπτυσσόμενος τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Περιορίζονται και σφαγιάζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίε. Τα μέτρα που προτείνονται πραγματικά είναι τρομερά ένα γιγαντιαίο σύστημα παρακολούθησης των πάντων. Αλήθεια, ποιον φοβάστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάστε τους λαούς. Γιατί φακελώνετε τους πάντες. Γιατί χρησιμοποιείτε τέτοιες βάσεις προσωπικών δεδομένων. Τρίτο, κοινο, ε, ε, κοινοτικοποίηση του ποινικού δικαίου. Καταργείται κάθε έννοια κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών. Και αυτό οι λαοί δεν δέχονται ούτε και πρόκειται να το δεχτούν. Τέλος, επειδή δεν έχουμε χρόνο κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι ο χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης χτίζει ένα θεσμικό πλαίσιο και μηχανισμούς για να διασφαλίσει αυτή την αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική που ζουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση λοιπόν των ίδιων των λαών είναι να απειθαρχήσουν, να μην υπακούσουν, να αγωνιστούν για να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ευχαριστώ. Πιέρ Λεγγιέ από την Εθνική Συνέλευση της Γαλλίας. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι υποστηρίζω 100% το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη και θα ήθελα να συγχαρώ τη Σουηδική Προεδρία καθώ και τον Επίτροπο Ζακ Μπαγό. Θα ήθελα να πω ότι άκουσα εδώ και εκεί σε διάφορε συνεδριάσεις Ε, να υπάρχει μια αντιπαράθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ θέλω να πω το αντίθετο, ότι είναι ένα τομέα και είμαι εθνικό βουλευτή, θα πρέπει τα εθνικά ε, κοινοβούλια και το, Εθνικό, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστούν πραγματικά στενά. Γιατί εξαρτάται από αυτό ε, η ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και η δημοτικότητα τη Ευρώπη. Όταν μιλάμε για αναρμόνιση των κανόνων, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, όταν μιλάμε για δικαστική συνεργασία, ε, στο αστικό δίκαιο, για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτά τα θέματα αφορούν όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως, αντί να φέρνουμε αντιμέτωπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αντίθετα θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και εγώ δεν σοκάρομαι, αντίθετα με διάφορους άλλους που μίλησαν πριν, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρξει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ ημών και ημών και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την κοινωτική πολιτική ασύλου πρέπει να πάμε πιο μακριά. Σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των παιδιών και γυναικών εναντίον τη εξεξουαλική εκμετάλλευση. Πρέπει να πάμε πιο μακριά. Σε ό,τι αφορά το Europol και τη Eurojust, πρέπει να πάμε πιο μακριά. Σε ό,τι αφορά το, Euro, ε, το Frontex, ε, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το Schengen αν δεν ενδυναμωθεί το Frontex. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ε, προσυπογράφω το πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει αυξημένες εξουσίες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και αυτό που χρειάζεται είναι μια θαυμάσια συνεργασία. Όχι μόνο για τα θέματα της επικουρικότητας, αλλά για όλα τα θέματα, για όλα τα ουσιαστικά θέματα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Τάβαρες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, um Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως απομακρύνομαι λίγο από το θέμα. Αλλά παρόλα αυτά σέβομαι τον ουσιαστικό τίτλο. Οικοδόμηση μιας Ευρώπης των πολιτών. Νομίζω ότι είναι μια σπάνια ευκαιρία ε, να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια. Φυσικά μπορούμε να μιλάμε για την Europol, την Eurojust, ε, τη Frontex για διάφορα θέματα. Για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την παρακολούθηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας, αλλά παρόλα αυτά δεν μιλάμε ακόμα για την Ευρώπη των πολιτών. Νομίζω ότι βουλιάζουμε σε μικροθέματα και μικροκείμενα ε, και, μικροκείμενα και ε, αποτυχάνουμε στις μεγάλες προκλήσεις, στα μεγάλα κείμενα, στα μεγάλα ζητήματα ασχολούμαστε με, πιο εύκολα με αγκουράκια, αλλά πολύ πιο δύσκολα ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το βάρος μιας συνταγματικής συνθήκης. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου εκλεγμένο σε μόνιμη βάση. Πρέπει να συνεργαστούμε για όλα αυτά στο διεθνή τύπο γίνεται λόγος για τη μελλοντική Προεδρία της Ευρώπης που θα επιλεγεί με βάση το αν την, τον θέλει το συγκεκριμένο άνθρωπο ο κ. Σαρκοζή ή η κυρία Μέρκελ. Δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια να δουν τι άτομο θέλουν οι χώρες τους να πάρει το θόκο του, της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά άτομο σημαίνει άντρα ή γυναίκα. Πέρα από αυτά που είπε ο Κάρλος Κοέγιο, ε, την ευθύνη που έχουμε, την, τη συνεργασία, υπάρχει και μια άλλη δοκιμασία, ότι πρέπει να είμαστε απλοί και να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να μιλήσουμε στους πολίτες μας ή απλώς κάνουμε νόμους για αυτούς ε, που τους επηρεάζουν μεν, αλλά δεν τους συμβουλευόμαστε δε. Όπως είπε και ο Ζίγμουν Μπάουμαν, θα πρέπει να είμαστε κάτι παραπάνω από νομοθέτε τώρα. Θα πρέπει να είμαστε και ερμηνευτέ των βουλών και θελήσεων των πολιτών μα. Αν περάσουμε στι μικρέ δοκιμασίε και χάσουμε τι μεγάλε, νομίζω δεν θα υλοποιήσουμε τον ε, στόχο μα. Ο κύριο Σκόφ από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξουν ένα πιο ένεργο ρόλο θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή συνεργασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Νομίζω ότι τα, οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να περιοριστούν στο να βρεθεί ο μικρότερος κοινό παρανομαστής. Για διάφορα μέτρα. Θα πρέπει βεβαίως να περιορίσουμε την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την εμπορία των ανθρώπων, την Ισλαμοποίηση, να εξασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή η ασφάλεια δεν είναι εξασφαλισμένη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό το σφαιρικό πρόγραμμα τιμώ και χαιρετίζω αυτούς που το κατήρτισαν. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν κάπου πηγαίνει λίγο πιο μακριά. Ίσως είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν, γιατί μπορούν να τεθούν προβλήματα. Υπάρχουν όρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Επίσης πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας και, τις, και το γεγονός ότι η προστασία και η ασφάλεια αφορά τον ίδιο το λαό μιας χώρας. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να λάβει υπόψη το αίσθημα που υπάρχει σε κάθε χώρα, ε, τότε νομίζω ότι θα έχει ε, περάσει αυτές τις δοκιμασίες και θα διασκεδάσει όλες τους τιμητές του. Ε, Νίτα από την Ρουμανική Βουλή. Ο κύριος Νίτα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα ακούσαμε τους ε, προλαλήσατε να αναφέρονται σε διάφορα σημαντικά θέματα. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ιδιαίτερος. Έχοντα υπόψη την ανάγκη να προστατεύσουμε και να προαγάγουμε τα δικαιώματα των πολιτών, δεν πρέπει να λησμονούμε και την ε, υποχρέωση να προαγάγουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Γιατί εδώ πρόκειται για μια ιδιάζουσα κατηγορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πρέπει ιδιαίτερη σημασία να αποδώσουμε, να αναγνωρίσουμε στα δικαιώματα των παιδιών. Ιδιαίτερα δε θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό υπό το πρίσμα της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης των πολιτών στα 27 κράτη-μέλη. Χρειάζεται ως εκ τούτου ένα συνεπές πλαίσιο μέτρων για τα, που, αφορά τα παιδιά οικογενειών που μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός παρακολούθησης έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων παιδιών, των παιδιών που βρίσκονται σε συνθήκες ε, φτώχειας γιατί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν ε, προσκόμματα βέβαια στην ανάπτυξη του παιδιού και θα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε περίπτωση διάκρισης εις βάρος των παιδιών. Ευχαριστώ και τώρα παρακαλώ τελευταίος ομιλητής, η τελευταία ομιλήτρια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ναι, όντως, η εναρμόνιση των δικαιωτικών χρόνων θα πρέπει να ξεκινήσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να καθοριστεί ξεκάθαρα σε ποια βάση θα γίνει αυτή η εναρμόνιση. Και αυτό από το έγγραφο που μας έχετε υποβάλει δεν είναι σαφές. Εμεί, ιδιαίτερα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι στα θέματα αυτά έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα και δεύτερον ότι δεν θα πρέπει να προκύψει υποβάθμιση των δικαιωμάτων για τα κράτη εκείνη τα οποία έχουν προχωρήσει περισσότερο. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία λοιπόν, ένα ελάχιστο προνομαστή. Επίση, υπόθηκαν πολλά για την Ευρώπη των πολιτών. Ελπίζω να υπάρξει μια μέρα και μια Ευρώπη των μεταναστών που έχει τεράστια σημασία, για την οποία όμως δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Και ρωτώ γιατί δεν υπάρχει στρατηγική στις προτάσεις, τις πολυάριθμες προτάσεις αυτού του εγγράφου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα περσινά ξινά στα φίλια που επαναλαμβάνονται και ξαναβλέπουμε διαρκώ και διαρκώ σε όλα τα κείμενα ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η λαθρομετανάστευση. Ε, όχι λοιπόν, πρέπει να βρούμε διαφορετικέ λύσει και προτάσει. Τον μιλούμε για φρόνταξη και για διεύρυνση των εξουσιών τη. Βεβαίω και θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα αναπτύσσει το πεδίο αυτό με γνώμονα την σύμβαση για τους πρόσφυγες της Γενέβης η οποία όμω δυστυχώ απουσιάζει από το κείμενο αυτό. Δεν έχει αναφερθεί στο κείμενο αυτό και θα θέλαμε κάποια ουσιαστικά νομοθετικά ε, βήματα προ τον ε, δρόμο αυτό προ τη λύση αυτή. Και ναι, πρέπει να υπάρχει μια κοινή στρατηγική, συμφωνώ και εγώ, αλλά το ερώτημα είναι πάντοτε το ερώτημα τη αναλογικότητα. Όταν μιλούμε λοιπόν για στρατηγική, για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, δεν βλέπω κανένα, καμία αιτιολόγηση η οποία να επιτρέπει στον αγώνα αυτόν να ποδοπατιούνται τα δικαιώματα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των πολιτών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, πράγματα στα οποία έχουμε δει τεράστιε παραβιάσει τον τελευταίο καιρό. Με το πρόγραμμα λοιπόν τη Στοκχόλμη δεν ξέρω αν μπορούμε να επιτύχουμε μερικά πράγματα. Φοβάμαι ότι δυστυχώ θα είναι πολύ κακά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ Όλου του ομιλητέ. Σχεδόν τηρήσαμε και το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μπούζεκ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συμπρόεδρε. Κάποιες, κάποια ενημερωτικά στοιχεία σημαντικά για όλους μας. Έχουμε τρεις ομάδες εργασίας. Η πρώτη ομάδα εργασίας, προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών και της Ευρώπης των δικαιωμάτων και των αξιών. Στην αίθουσα, εδώ, που είσαστε τώρα, εδώ στο κύκλιο. Η δεύτερη ομάδα εργασίας, μια Ευρώπη της δικαιοσύνης, της δημοκρατικής λογοδοσίας και της ασφάλειας δικαίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην απέναντι αίθουσα, στον ίδιο όροφο, τρίτο όροφο δηλαδή, είναι η αίθουσα με νούμερο 3C50, απέναντι ακριβώς από την αίθουσα που βρίσκεστε. Και η τρίτη ομάδα εργασίας, προστασία των πολιτών ευρωπαϊκός ε, χώρος, εσωτερικός ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας. Πού θα συναντηθείτε δύο ορόφους κάτω από εδώ που βρισκόμαστε, στον πρώτο όροφο δηλαδή. Η αίθουσα έχει νούμερο 1α002, στο ίδιο κτίριο που βρισκόμαστε τώρα. Υπάρχουν βέλη για τις αίθουσες συνεδριάσεων και έχετε επίσης την πληροφορία και στα, στους φακέλους σας. Οι εισηγητέ των τριών ομάδων εργασίας θα παρουσιάσουν τις εκθέσεις κατά προτίμηση γραπτών, είτε γαλλικά είτε αγγλικά, γιατί αγγλικά και γαλλικά αποφασίστηκε ότι είναι οι γλώσσες εργασίας μας. Αύριο στην Ολομέλεια το πρωί θα παρουσιαστούν όλες οι εκθέσεις και στις 7 και 4 σήμερα το βράδυ θα παραθεθεί επίσημο δείπνο. Θα ήθελα να καλέσω όλους σας στις 7 και 4 το απόγευμα για το επίσημο δείπνο στο ιδιωτικό εστιατόριο των ε, βουλευτών. Είναι ένα κτίριο στα αριστερά σας, βγαίνοντας από εδώ, στρίβετε αριστερά και επίσης υπάρχουν βέλη για να φτάσετε ως το εστιατόριο. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε σήμερα το, απόγευμα, το βράδυ δηλαδή και αύριο το πρωί. πέρα από τις σημερινές ομάδες εργασίας, θα ήθελα αύριο το πρωί στις 9.30 να είστε όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε την Ολομέλεια. Λοιπόν, αυτά από, από μας τους δύο προέδρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, έχουμε και τις σημερινές ε, ομάδες εργασίας και φυσικά το επίσημο δείπνο. Γεια σας.